στήριξη της εμπορικής πολιτικής. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε και την αντιμετώπιση των εμπορικών θεμάτων και όχι να συζητάμε όλα τα άλλα εκτός από το εμπόριο. Ευχαριστώ κύριε Κασπάρη. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Άσενς, για ένα, για ένα λεπτό.